επί του θέματος. Αυτό είναι ο μόνο, το μόνο νομικό πλαίσιο για να προχωρήσουμε. Έληξε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο σημείο σε διάταξη είναι η κοινή συζήτηση σχετικά με την αλληλεία. Η σύσταση του κυρίου Βαλέσα, τη Σύμβαση περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλληλείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού και η έκθεση της κυρίας Φράγκα Εστέβες, σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλίας στο βορειοανατολικό Ατλαντικό. θα τηρώ πολύ αυστηρά του, τα χρονικά διαγράμματα για όλους τους ομιλητές. Ε, παρακαλώ για την κατανόησή σας. πρώτος έχει το λόγο ο εισηγητής, ο κύριος Βαλέσα, για τέσσερα λεπτά. panie κύριε πρόεδρε κύριε επίτροπε αγαπητοί συνάδελφοι η συνθήκη που θα σας παρουσιάσω ξεκίνησε να υπογράφεται το 1978 στην Οτάβα και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1979. Ουσιαστικά συνέστησε την οργάνωση Αλίας Βορειοδυτικού Ατλαντικού για να μεγιστοποιήσει την χρήση και να διαχειριστεί ε, ορθολογιστικά τους αλλιευτικούς σπόρους. Τροποποιήσεις έγιναν το 2007 και το 2008. Ενώ αυτό το έγγραφο εισάγει σημαντικές μεταβολές, δηλαδή εναρμονίζεται η σύμβαση αυτή με άλλες συμβάσεις περιφοριακού χαρακτήρα, καθώς και με άλλους μηχανισμούς διεθνείς. Έλεγα λοιπόν ότι η οργάνωση και η δομή της οργάνωσης εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει σαφής κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ κρατών σημαίας, κρατών λιμένα και συμβαλωμένων μερών. Η διαδικασία είναι ομαλή πλέον, καθώς και ο προϋπολογισμός και υπάρχουν μηχανισμοί επίλυσης διαμάχης που έχουν θεσπιστεί. Λοιπόν, σε σχέση με αυτή τη σύμβαση και την έγκριση αυτών των τροποποιήσεων θα έλεγα ότι είναι προς όφελος όλα αυτά προς όφελος ΕΕ. Λοιπόν, αξίζει να την υποστηρίξουμε. Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα όσον αφορά τη διαδικασία έγκρισης. Πρώτον, τα συμβαλόμενα μέρη υιοθέτησαν τροπολογίες το 2007 στα αγγλικά. Το 2008 εκδόθηκαν οι τροποποιήσεις, το στα γαλλικά. Όσον αφορά τώρα τη μεταγραφή σε ευρωπαϊκό δίκαιο, φτάσαμε στο 2010. Αυτό σημαίνει ότι για να εξελιχθεί αυτό το έγγραφο στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάστηκαν δύο χρόνια. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε μια τέτοια καθυστέρηση. Η άμεση ανταπόκριση είναι κλειδί στις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, το το Κοινοβούλιο πρέπει να βρει τρόπους να αποφύγει την επιβράδυνση των δικασιών και σύμφωνα με τη Λισαβόνα πρέπει να επισπεύσουμε την διαδικασία λήψη αποφάσεων. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε διαπιστώσει τα πράγματα δεν πάνε ομαλά και πρέπει να ενεργήσουμε. Θα ήθελα ακόμη να σας πω ότι τον Δεκέμβριο του 2009 τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Ωραία. Η Επιτροπή Αλίας τώρα πρέπει να εκπροσωπείται όπως και το Κοινοβούλιο πρέπει να εκπροσωπείται παρκώς στην διαπραγμάτευση τέτοιων συμβάσεων. Το 2007 και 2008 το Ευρωκοινοβούλιο δεν εκπροσωπήθηκε με αυτόν τον τρόπο για προφανείς λόγους. Μπορούμε βεβαίω να εγκρίνουμε μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, αλλά θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στο Συμβούλιο και στην Κομισιό ότι πρέπει να σέβονται τις νέες αρμοδιότητες μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψατε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη προ το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί φτάσαμε, καταλήξαμε σε αυτή την καλή συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση και ιδιαίτερω στι νομικέ υπηρεσίε των τριών θεσμικών οργάνων για την συνεργασία και τη βοήθειά του προκειμένου να επιληθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη νέα διαδικασία επιτροπολογία απολογίε συνθήκη τη Λισαβόνα. Νομίζω ότι πετύχαμε ένα καλό συμβασμό, γιατί σημαίνει μια σημαντική πρόοδο εν σχέση με την παρούσα κατάσταση, παρόλο που όλοι βεβαίω χρειάστηκε να κάνουμε κάποιες παραχωρήσεις στα πλαίσια μιας ιδιαίτερως πολύπλοκης εργασία, Μια και η πρόταση της Επιτροπής ε, μας ε, έθεσε πρώτη ημερομηνία σε θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνα. προκειμένου το να ε, εφαρμόσουμε το άρθρο 291 όσον αφορά τις εκταλιστικές πράξεις και τις καταξιδότηση πράξεις όσον αφορά τις συστάσεις που προέρχονται από τις περιφερικές οργανώσεις της Αλίας. Ο σκοπός του Κοινοβουλίου ήταν βασικά να θεσπίσει έναν μηχανισμό που να επιτρέπει να προβούμε σε αυτή τη μεταγραφή στο με το ταχύτερο τρόπο. Να, να αποφύγουμε επίσης τους ε, διάφορους γραφειοκρατικούς γραφειοκρατικούς φραγμούς. Η νέα σύνταξη του άρθρου 48 που αφορά το συμβιβασμό που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο σε σχέση με τις προηγούμενες τροποποίησεις αυτού του κανονισμού θα επιτρέψει στην Επιτροπή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις, υποχρεώσεις και να ε, διατυπώσει νέες ε, συστάσεις. Είναι βέβαιο ότι η Επιτροπή θα ήθελε όλα τα άρθρα της πρότασης να μπορούν να αναθεωρηθούν μέσω των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Ενώ η συμβαστική και η συμβαστική λύση το αποδέχεται όσον αφορά τις μεταφορτώσεις και τις περιπτώσεις παραβίασης καθώς και τα τάκ, δηλαδή θέματα τα οποία σχετίζονται σε θέματα ελέγχου στο πλαίσιο αυτής της ε, συναπόφασης. Το Κοινοβούλιο δεσμεύεται να τροποποιήσει, κυρία Επίτροπη, αυτή την, αυτό τον κανονισμό εάν αποδειχθεί ότι στο πλαίσιο της συναπόφασης είναι δυνατόν να τεθούν σε αμφισβήτηση ή σε κίνδυνο οι υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως συμβαλόμενου μέρους της, των περιφερειακών οργανώσεων της Αλίας. Γι' αυτό θεωρούμε ο συμβασμός αυτός είναι μια σημαντική πρόοδος όχι μόνο όσον αφορά αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση αλλά όσον αφορά τις βάσεις μιας μελλοντική συζήτησης μεταξύ Επιτροπής, Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όσον αφορά την ελευθερική πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εξ Επιτροπής, ε, η κυρία Δαμανάκη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, the Commission urges η Επιτροπή παρακαλεί το Ευρωκοινοβούλιο να εγκρίνει τι τροποποιήσει της ε, οργάνωση αλληλείας βορειοδυτικού Ατλαντικού, τρόπολογίε δηλαδή για τη Σύμβαση ΝΑΤΟ. ΝΑΦΟ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ και τον κύριο Βαλέσα για τη βοήθειά του. Αυτή η τροπολογία τροποποιεί τη σύμβαση για να γραμμιστεί με άλλες περιφερειακές συμβάσεις και διεθνείς μηχανισμούς λαμβάνει υπόψη του την ευθυγράμμιση της αλίας και προσδιορίζει τις ευθύνες των κρατών σημαίας, κρατών λιμένα και προσδιορίζει και τον μηχανισμό λήψης απόφασης. Εξυγχρονίζει το προϋπολογισμό και προσδιορίζει ακόμη τον, την επίλυση των διαφορών. Αυτές οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, πραγματοποιήσει της υποχρεώσει της, της διεθνής όσον αφορά την αλλία. Χρειάζεται επίσπευση της έγκρισης των τροπολογιών προς συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας παρακαλώ να βοηθήσετε. Και τώρα αναφέρομαι στην δεύτερη έκθεση που αφορά τη Σύμβαση Συνεργασίας στη Βόρειο-Ανατολική στο βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό πάντα για την Αλία. Ευχαριστώ την κυρία Φράγκα για την έκθεσή της. Χαίρομαι που έχουμε υποστήριξη της Επιτροπής Αλίας σε σχέση με αυτή την πρόταση. Η εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στην ΕΑΦΚ σίγουρα θα μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε την αλία στην Ατλαντική περιοχή. Ε, όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Κομισιόν δεν είναι τελείως ικανοποιημένη με το πακέτο που συμφωνήθηκε μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου κατά το τρίλογο με την Κομισιόν. Έχω απογοητευτεί από ορισμένα αποτελέσματα, ειδικότερα όσον αφορά το άρθρο 48 που έχει να κάνει με τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού. Η Κομισιόν ήθελε περισσότερη εκχώρηση εξουσίες για τη μεταγραφή τροπολογιών. Μελλοντικά αυτό. Θα ήθελα να σας εξηγήσω γιατί και σας παρακαλώ προσέξτε δε, γιατί θα έχουμε και μελλοντικά τα ίδια προβλήματα. Ως, πώς γνωρίζετε, πρέπει να εφαρμόσουμε πλήρως το ΣΥΜ γιατί είναι υποχρέωσή μας διεθνής βάσει της συνθήκης ΝΕΑΦΚ. Σύμφωνα με αυτή τη συνθήκη, οι τροπολογίες γίνονται ε, δεσμευτικές 80 μέρες μετά την υιοθέτησή τους. 80 μέρες λοιπόν έχουμε. Πραγματικά ανησυχώ που οι ε, περιορισμένες εξουσίες που έχουν εκχωρηθεί στην Κομισιόν μπορεί να παρεμποδίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή. Και αυτή είναι η πραγματικότητα και μια απάντηση προς τον κύριο Βαλέσα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Αυτή όμως δεν είναι δικιά μου ευθύνη. Θέλω όμως να συνειδητοποιήσετε τα γεγονότα. Πρέπει να αποφύγουμε τη μεταφορά μέτρων ΝΕΑΦΚ σε μύθο του Σισίφου σήμερα. Τα μέτρα του περασμένου έτους της ΝΕΑΦΚ μεταγράφονται τελικά όταν υιοθετηθεί το πακέτο. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα η ΝΕΑΦ θα υιοθετήσει νέα μέτρα. Πράγμα το οποίο θα σημαίνει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχές 2011. Λοιπόν, γι' αυτό ο κανονισμός αυτός δεν προκαταλαμβάνει τη θέση μας όσον αφορά την χρήση των άρθρων 290 και 291 της συνθήκης σε σχέση με την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταγραφή των διατάξεων για την περιφερειακή αλληλεία. Επίσης, η Κομισιό επιφυλάσσεται το δικαίωμά της να προτείνει τροποποιήσεις καθώς και αποφάσεις εφαρμογής. Εάν η μεταγραφή σύμφωνα με την νομοθετική διαδικασία ε, οδηγήσει σε καθυστερήσεις, ε, τότε υπονομεύεται το καθήκον μας να συμμορφωθούμε με διεθνείς υποχρεώσεις και θα ενεργοποιηθούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φράγκα και τον κύριο Βαλέσα για τις εκθέσεις τους και την Επιτροπή Ελίας για τη δουλειά που έκανε πάνω σε αυτό το θέμα. Τώρα πρώτος ο κύριος Καντέκ για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Δαμανάκη, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να μιλήσω για την έκθεση Φράγα κυρίως. Είναι ύψης της σημασίας για την ενίσχυση των ελέγχων στο βορειοανατολικό Ατλαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι από κοινού νομοθέτης σε θέματα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Είναι μία από τις προτεραιότητές μας να καταπολεμήσουμε τη μη ρυθμισμένη και μη δηλωμένη αλία που δημιουργεί δυσχέρειες για τους δικούς μας αλληλείς. Πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό και παραοικονομία, διότι οι πλειοκτήτες οι οποίοι είναι παράνομοι δεν τηρούν το δίκαιο της θάλασσας και καταβάλουν χαμηλά η ημερομίσθια στους εργαζόμενους. Ο κανονισμός INN μιλά για κόστος εργασίας το οποίο δεν είναι πια ανταγωνιστικό για τους Ευρωπαίους πλειοκτήτες. Γι' αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε ανωδική πορεία ως προς τους μισθούς και τα σχετικά. Υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει διαχείριση και ρύθμιση καθώς και έλεγχος έτσι ώστε να έχουμε αηφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αλίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παρακολύονται οι αλληλεί στο έργο τους. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε με κυρώσει την παράνομη αλία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την πρόεδρό μας για αυτή την έκθεση και πιστεύω ότι το ΣΕΠΑΝ θα πρέπει να ισχύσει στο ευρωπαϊκό δίκαιο και θα πρέπει και οι μη συμβαλόμενοι να τηρήσουν αυτό, αυτές τις διατάξεις. Επίσης, σε σχέση με το άρθρο 290 της ε, κατεξιοδότηση πράξης, θα πρέπει να τηρηθεί αυτό το άρθρο, καθώς και η κατεξιοδότηση πράξης στο παράρτημα και να διατηρήσουμε μία θεσμική ισορροπία. Εμείς ως από κοινού νομοθέτης θα πρέπει να έχουμε πλήρη ελευθερία για τι ε, κατεξουσιοδότηση πράξη. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε, κυρία Δαμανάκη, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που μπορούμε να αποφασίσουμε ένα κανονισμό που συνιστά ένα παραπέρα βήμα στον κοινό μας δρόμο προς μια βιώσιμη αλεία. Οι περιφερειακές οργανώσεις αλείας είναι εξαιρετικά σημαντικές για μια καλή διαχείριση σε παγκόσμια κλίμακα. Δυστυχώς οι διαπραγματεύσεις συχνά είναι δυσχερείς και για κάποιου ανυπόμενου ανθρώπου όπω είμαι εγώ, εξαιρετικά βραδίε. Γι' αυτό θα πρέπει να πράξουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ούτω ώστε οι περιφερειακές οργανώσεις αλλία να ενισχυθούν. Όσον αφορά το, την έκθεση αυτή τη ε, ΝΕΑΦΣΑ, θα ήθελα να πω ότι οι νέοι έλεγχοι για τα κράτη λιμένος και τα νέα μέτρα για την ε, παρεμπόδιση της παράνομης αλίας είναι ευκταία μέτρα. Παρ' όλα αυτά ε, έπρεπε να διαπραγματευτούμε σκληρά με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για θέματα που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν τεχνικής φύσεως, παρόλα αυτά είναι σημαντικά για το μελλοντικό μας έργο. Θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να... βρήκαμε ένα σωστό συμβασμό όσον αφορά τη κατεξοδότηση πράξης επίσης για το θέμα το πώς οι μελλοντικές αποφάσεις της ΝΕΑΦΣ θα μεταγραφούν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Δεν είναι μυστικό ότι η Επιτροπή όμως δεν είναι ιδιαίτερως ευτυχής με το αποτέλεσμα και μπορώ να το κατανοήσω, γιατί δεν πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόσει τις αποφάσεις της ΝΕΑΦΣ. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποδείξουν από κοινού ότι εκεί όπου παρίσταται ανάγκη είναι σε θέση να ολοκληρώσουν μια διαδικασία συναπόφασης γρήγορα. Τέλος, για το θέμα αυτό την ε, αντιπαράθεση με τις χώρες Μακρέπ όσον αφορά τα διεθνή ύδατα για τον ε, νοτιοανατολικό Ατλαντικό. Ε, χρειαζόμαστε μία συμφωνία για ίδιο όπως είναι τα σκουμπριά. Και ξέρετε ότι δεν έχει επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Θεωρώ ότι είναι τετέρως λιβερό παρά την ε, εύρυθμη, παρά την καλή συνεργασία ότι υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Ε, θα έπρεπε ίσως να δώσουμε στις περιφερειακές οργανώσεις ε, αλλίες αρμοδιότητες για τα, περιφερειακά για τα μεταναστευτικά είδη όσον αφορά την παράκτια αλλία. Νομίζω ότι θα ήταν ριζοσπαστικό αυτό το μέτρο, αλλά επιθυμητό. Η κυρία Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι με την ε, συμφωνία για την μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλίας στον ε, βορειοδυτικό Ατλαντικό δημιουργήθηκε μια πολύ σημαντική οργάνωση. Σκοπός της είναι η διατήρηση και η βέλτιστη χρησιμοποίηση των αλληλευτικών αποθεμάτων στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό. Η σύμβαση αυτή, η συμφωνία, τροποποιήθηκε στη συνέχεια και προσαρμόστηκε σε άλλες περιφερειακές συμβάσεις. Σύγχρονα μοντέλα διαχείρισης των αποθεμάτων υιοθετήθηκαν σε αυτή την τροποποιημένη σύμβαση. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό η δομή του οργανισμού να είναι πιο αυστηρή και να είναι ξεκάθαρα ορισμένε οι αρμοδιότητες των συμβαλόμενων μερών. Επίσης θα ήταν ευταίο να υπάρχει δυνατότητα επίλυσης των διαφορών μέσω ενός μηχανισμού διαιτησίες οι διαφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματικά παρουσιάζουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Το Κοινοβούλιο θα έπρεπε στο πλαίσιο των νέων του αρμοδιοτήτων που στηρίζονται στην, ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας να δώσει τη συγκατάθεσή του. Ως και όδηση συγγήτρια της Άλντε, εγώ είμαι υπέρ της τοποθέτηση ε, ε, τοποθέτησης του κυρίου Βαλένσα. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λόβιν για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Επίτροπε, μέλη του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φράγκα και τον κύριο Βαλανίσκα για τις εκθέσεις που συζητάμε σήμερα. Η Επιτροπή αυτή είναι πολύ σημαντική, ο ΝΑΦΟ δηλαδή και η ΝΕΑΦΚ είναι πολύ σημαντική για την Ευρώπη και γενικά είναι θετική μεταρρύθμιση, πράγμα το οποίο δεν σημαίνει πάντοτε για την ΑΠΟ. Αν και η ΝΙΑΦ καποδίδει καλύτερα από άλλες περιπτώσεις, η κατάσταση των αλλιευμάτων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους η απόδοση δεν μπορεί να αξιολογηθεί και αυτό συνεπάγεται ότι υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες κατά πόσο οι συνθήκες για τη βέλτιστη ε, εκμετάλλευση έχουν υλοποιηθεί. Έχει βελτιωθεί όμως η εποπτεία, η παρακολούθηση και η εφαρμογή μαύρης λίστας και αυτά οπωσδήποτε είναι μεγάλα επιτεύγματα. Από την αξιολόγηση βλέπουμε ότι υπάρχει και ένας μηχανισμός ε, επίλυσης ε, διαφωνιών, αλλά η μεταγραφή αυτών των μέτρων πήρε πάρα πολύ χρόνο από την Κομισιόν το 2007 υιοθετήθηκαν, φτάσαμε στο 2010. Θα πρέπει δηλαδή να αναλάβουμε και τις διεθνείς μας ευθύνες πιο γρήγορα. Η καταπολέμηση της παράνομης αλληλεία είναι πολύ σημαντική. Περίπου 30% των αλλιευμάτων είναι παράνομα. 11 με 12 εκατομμύρια τόνοι ψαριών, 23 δις ε, ευρώ δηλαδή, εκφορτώνονται παράνομα. Είναι ένα πέμπτο του, των επίσημων αλλιευμάτων. Θέλουμε λοιπόν βιώσιμη εκμετάλλευση των αλλιευμάτων και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Η εφαρμογή του κανονισμού είναι πολύ σημαντικός μηχανισμός και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλληλείς προσπαθούν να αλλάζουν χώρους αλίευσης, ε, κράτη σημαίας, κράτη λιμένων και όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε προβλήματα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Οι μηχανισμοί συμμόρφωσης μπορεί να συνεπάγονται μεταβολή περιοχών αλίευσης και μεταβολή ε, κρατών σημαίας. Το λέμε δε αυτό flag hopping. Και χρειαζόμαστε να έχουμε περισσότερη συνεργασία βεβαίως. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να δημιουργήσουμε ένα συνολικό μητρό αλλιευτικών ε, πλοίων ε, που να καταδεικνύουν με σαφήνεια τον ιδιοκτήτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει την αλία με υπευθυνότητα. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση που τονίζει το θέμα του ελέγχου και της επιθεώρησης. Επειδή μιλάμε για κοινοτικά ύδατα, ε, υπάρχουν τομείς που δεν τη χάνουν ελέγχου και επιθεώρησης. Θα πρέπει να καλύψουμε όλα τα κοινοτικά ύδατα, τα κοινοτικά ύδατα στο σύνολό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν υπάρχει ένας και μοναδικός τρόπος ε, κατανομής ποσοστώσεων και κοινοποίησης αλλιευμάτων των ε, κρατών μελών. Από ό,τι φαίνεται, η Επιτροπή δεν έχει λάβει γνώση. Και πολλές φορές οι γνωμοδοτήσεις Επιτροπής είναι αντιφατικές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη του, τον πληθυσμό ρεγκών στο, στη Βαλτική θάλασσα διότι από το 2004 έχουμε ε, εξετάσει τα αίτια αυτής της κατάστασης, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε μία λογική εξήγηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει βεβαίως είναι και το ηχθιέλεο και τα ηχθιάλευρα. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο ο φορέας επιθεώρησης και ελέγχου είναι επιλεκτικός όπως ισχύει για την Ανατολική Βαλτική. Επίσης, τα σκάφη ε, βιομηχανικής αλίας την χάνουν άλλες, ε, άλλες μεταχείρισεις και πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη και το North Stream και κατά πόσο από εκεί υπάρχει απώλεια εσόδων. Όλα αυτά θα πρέπει να μας απασχολήσουν μεμονωμένα. Ευχαριστώ. Um, Mr. President. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε Δαμανάκη. Πράγματι είναι βεβαρημένη η εργασία απόψε. Έχουμε συναντηθεί ήδη στην Επιτροπή Αλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές για αυτές τις εκθέσεις και να επαναλάβω το σχολείο πολλών συναδέλφων εδώ σε σχέση με την ανησυχία τους για την καθυστέρηση στην πρόοδο και την εξέλιξη αυτών των υποθέσεων. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να μιλήσω για τις αλλιευτικές συμφωνίες γενικότερα και να τονίσω την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ όλων των συμβαλωμένων μερών. Αυτό αναφέρθηκε ήδη από την Επίτροπο όταν είπε ότι οι συμφωνίες συμνεπάγονται μεγαλύτερη ευθύνη από όλους τους εμπλεκόμενους. Για φανταστείτε ότι έχετε κάνει μια τεράστια επένδυση ε, σε, σε ένα εργοστάσιο που, έχει, που παράγει ένα προϊόν από ανανεώσιμη πηγή σε υψηλότατο ποιοτικό επίπεδο και τότε ο γείτονα σα αποφασίζει να σκίσει τη Διεθνή Συμφωνία και να δηλώσει ότι επεκτείνει μαζικά το μερίδιο του από τους φυσικούς πόρους από το οποίο εξαρτάται η επιχείρησή σας. Αυτό συνέβη με, τη, με το σκουμπρί και ειδικότερα με μια επιχείρηση στην Βόρεια Ιρλανδία. Αναφέρομαι στην συμφωνία μεταξύ Φερών, Ισλανδίας κτλ. Ακούσαμε την Επιτροπή και χαίρομαι για την ε, στεναρή θέση που έχετε υιοθετήσει κυρία Επίτροπε. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειές σας, αλλά θέλουμε να παροτρύνουμε την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο να σας στηρίξει προσπαθώντας όσο προσπαθείτε να διαπραγματευτείτε μία επίλυση σε μία πατηλή και δύσκολη κατάσταση. Για λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν τρεις ομιλητές από την Ιρλανδία απόψε, κυρία Ντότς, ο κύριος Μπόκ που θα μιλήσει και εγώ. Και μεταξύ των τριών μας εκπροσωπούμε όλη την αλληλευτική κοινωνία της Ιρλανδίας. Η αλληλεία είναι πολύ σημαντική στη χώρα μας για πολλά χρόνια. οι παράκτιες κοινότητες εξαρτώνται από αυτήν. Όπως είπα, Ποτέ δεν είχα απογοητευτεί περισσότερο ε, μιλώντας με τους αλλιείς λόγω της παράνομης αλλίας, της έλλειψης ιχνήσεων με συγχωρείτε δεν μπερδεύτηκα ε, και έχουμε και εισαγωγές ε, ψαριών αμφίβολης κατάστασης και ποιότητας. Οι εισηγητές ευτυχώ αναφέρονται σε αυτό το θέμα τα απόψη και χαίρομαι για την ε, ΝΑΕΦΣ η οποία προτείνει να εκφορτώνονται να μην εκφορτώνονται σε ευρωπαϊκά λιμάνια αλλιεύματα χωρίς την εποπτεία της χώρας σημαία της Ευρωπαϊκής. Και αυτό είναι πολύ σημαντική διαβεβαίωση για τις κοινωνίες μας ακόμη. Είναι πολύ σημαντικό για το Ευρωκοινοβούλιο να διατηρήσει το προνόμιό του, να εξετάζει μελλοντικέ τροποποιήσεις της σύμβασης αυτής. Εξίσου σημαντικό είναι η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να συνεργαστούν από κοντά ώστε να εξασφαλίσουν τα ωφελήματα που απαιτούνται για τις παράκτιες κοινότητες που είναι βασικά αλλιευτικές. Ακόμη δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία αυτή χωρίς να εξετάσουμε την ανάπτυξη της ηχθειοκαλλιέργειας. Είναι πολλά που μπορούμε να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μεγάλη ευκαιρία ακριβώς σε αυτή την οικονομική κρίση να αναπτύξουμε την ηχθειοκαλλιέργεια. Gracias, presidente. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρία Δαμανάκη και συγχαρητήρια στους δύο εισηγητές, τον κύριο Βαλέστα και την κυρία Φράγα. Η έκθεση αυτή της κυρίας ε, Φράγα είναι η έκθεση συνεπία των, ε, σε συνέχεια των συστάσεων της, που διατύπωσε η ΝΕΑΦ το 2006. Παρόλο που η σύμβαση ε, η Σύμβαση αναδιατυπώνει τα μέτρα ελέγχου στις ε, ζώνες της Σύμβασης. Η κυρία ε, Φράγα αναφέρεται στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι βασικές τροποποιήσεις είναι η εκπλήρωση των προδιαγραφών για τα μη συμβαλόμενα, εκ μέρους των μη συμβαλόμενων μερών και επίσης η ευθυγράμμιση με άλλες συμβάσεις, μέτρα διαχείρισης των λευτικών αποθεμάτων και νέα μέτρα κατά καταπολέμησης της παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που υπόθηκε προηγουμένως, τόσο στην έκθεση της κυρίας Φράγα που εγκρίθηκε το 2006, παρόλο που η σύμβαση ε, είχε ε, θεσπιστεί πολύ νωρίτερα θα ήθελα να εκφράσω την διαφωνία μου με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τη μεταγραφή των συστάσεων των περιφερειακών οργανώσεων αλίας. Όχι μόνο θα πρέπει να έχουμε μια παρακολούθηση της παράνομης αλίας μέσω των ποσοστώσεων και των ΤΑΚ, αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένας αγώνας κατά του νομικού κενού όσον αφορά την έλλειψη μεταγραφής των κανόνων δεν αρκούν οι συστάσεις άλλων κανονισμών γιατί ε, χρειάζεται περισσότερη αξιοπιστία. Επίσης αμφισβητείται τελικά η διαδικασία της συναπόφασης και η ισορροπία μεταξύ θεσμικών οργάνων. Θα πρέπει να εφαρμοστούν ε, το τάχιστο δυνατό τα μέτρα αυτά ε, και να δοθεί η σωστή προτεραιότητα στις περιφερειακές οργανώσεις αλίας. Το κοινοτικό δίκαιο η μη τήρηση του κοινωτικού δικαίου όσον αφορά τη μεταγραφή όλων αυτών των μέτρων που έχουν ληφθεί από τις περιφερειακές αργανώσεις είναι εις βάρος του Κοινοβουλίου και θέτει σε αμφισβήτηση τη συνθήκη της Λισαβόνας. Είπε η Επίτροπος ότι θα υπάρξουν νέες συμφωνίες αλλά ζητούμε από την Επιτροπή ταχύτητα όσον αφορά την νομική εφαρμογή. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα νομικό κενό ε, που δίνει πολλά περιθώρια στην παράνομη και λαθρέα αλία. Ε, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ και τους δύο εισηγητές για τις εκθέσεις και να αναφερθώ στην έκθεση Φράγα που δεν ε, ε, δημιούργησε διαφωνίες γιατί όλοι δεχτήκαμε το συμβιβασμό έτσι ώστε να έχουμε μακροχρόνια διατήρηση και ευέλτιστη ε, δυνατή χρήση των πόρων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να θίξω το θέμα της διαφωνίας που υπάρχει σε σχέση με το σκουμπρί και την αλία του στο βορειοανατολικό Ατλαντικό. Θα πρέπει το θέμα να επιληθεί το συντημότερο δυνατόν, διότι η υπεραλίευση θα έχει ολέθρια συνέπεια στα μελλοντικά αλλιεύματα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να το δεχτούν. Οι πρόσφατες συζητήσεις στο Λονδίνο δεν οδήγησαν πουθενά θα επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα. Εύχομαι κάθε επιτυχία και ελπίζω να επικρατήσει η λογική. Κύριε Επίτροπε, στις 26, μετά τις 26 θα αποτιμήσετε την κατάσταση και χαίρομαι για τη στεναρή σας τάση. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει αυτά τα αλλιεύματα να είναι και να παραμείνουν υγιή και για το μέλλον. Επίσης, δεν μπορούμε να επαναλαμβάνουμε τα σφάλματα του παρελθόντος σε σχέση με το προσφυγάκι. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να έχουμε ένα υγιές αλίευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάτσεν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω τις εκθέσεις που συζητούνται απόψε. Πρέπει να επίσης να υποφελθώ της ευκαιρίας για να κάνω ορισμένε γενικές παρατηρήσεις για τις διεθνείς και πολυμερείς συμφωνίες για την αλία αν οι συμφωνίες μεταξύ κρατών αλλιευτικών πρέπει να πετύχουν, πρέπει τα κίνητρα να είναι σαφή για όλα τα μέρη, ώστε να εφαρμόζονται τα μέτρα συντήρησης και διατήρησης. Ακόμη χρειαζόμαστε επιστημονική συμβουλή για την βάση, ώστε να αποτελέσει τη βάση των σχεδίων διαχείρισης και συντήρησης. Εκ μέρους της περιφέρειάς μου της Σκοτίας, η κοινή πολιτική αλληλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπήρξε μεγάλη επιτυχία. Το σχέδιο ουσιαστικά έχει οδηγήσει στην απόρριψη υγιών αλλιευμάτων και η σημερινή διαφωνία για το σκουμπρί, όπως ακούσαμε από άλλους ομιλητές, έχει μεγάλες επιπτώσεις για όλες τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Υπάρχει άραγε ελπίδα να επιτύχουμε καλές συμφωνίες μεταξύ αλλιευτικών κρατών χωρίς να απειλούνται τα αποθέματα προς εξαφάνιση στο τέλος. Μονομερός. Θα ήθελα η Επιτροπός να συνεχίσει ε, να αναζητεί μια λύση. Ξέρω ότι γνωρίζει τα συναισθήματα των σκότων. Επισκέφθηκε τη Σκοτία πρόσφατα. πρόσφατα. Θα ήθελα λοιπόν η Επίτροπος να έχει υπόψη της ότι έχουμε επιστημονικές σίγουρες σύμβουλες. Πρέπει τα σχέδια να είναι οργανωμένα και αποτελεσματικά και κυρίως πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για εκείνους που υπόκεινται σε αυτά τα σχέδια, δηλαδή για τις αλλιευτικές κοινότητες, ώστε να συμμορφούνται. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, η μη διευθετημένη αλληλεία καταστρέφει τις παράκτιες περιοχές και μπορεί να αποτελέσει απειλή για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Γι' αυτό χαιρετίζω αυτή τη συμφωνία με το Συμβούλιο και θεωρώ ότι έχει επιτευχθεί ένα περαιτέρω βήμα μέσα στα πλαίσια της ΝΑΦΟ. Η ενδυνάμωση και ενίσχυση μέτρων καθώς και μία ρωμαλαία νομοθεσία μπορούν να μας βοηθήσουν στην προστασία πόρων ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχει υπερεκμετάλλευση. Παρόλα αυτά, η εφαρμογή αυτού του κανονισμού δεν επιτρέπει την, την πλήρη αντιμετώπιση της παράνομης αλίας ή της μη ρυθμισμένης αλίας, γιατί ορισμένα κράτη-μέλη δεν θέλουν να εφαρμόσουν τις διεθνείς συμβάσεις. Γι' αυτό ε, πλήττονται οι θαλάσσιοι πόροι. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ε, οι συνθήκες εργασίας που αποτελούν μια μορφή δουλείας. Πρώτα ο κύριος ε, Σικέρσκι για ένα λεπτό. Mr. Sikorsky, for one minute, catch the eye. Szanowni Państwo, konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy. Κυρίες και κύριοι, οι συμβάσεις ως προς την ε, μελλοντική συνεργασία στο Βόρειο Ατλαντικό θα πρέπει να εναρμονιστούν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Μιλάμε για βέλτιστη χρήση των ε, υπαρχών των πόρων, επαρκή διαχείριση των ε, αλλιευτικών πόρων και μία συστημική προσέγγιση της αλίας. Επίσης, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλία. Όλες αυτές οι αλλαγές θα οδηγήσουν στη βιώσιμη αλληλεία, αλλά θα πρέπει να διαχειριστούμε και να επιτηρούμε την διαδικασία αυτή διαχρονικά, ως προς τα επίπεδα αλλιευμάτων δηλαδή, και να προσαρμόζουμε τις αποφάσεις μας. Για ένα λεπτό. <coughs> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τις ε, σχετικές συμφωνίες, ο επικεφαλής τη αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκε να εκχωρήσει στους ε, αλληλείς ε, του Σαν Νικολό τις γαλλικές ποσοστώσεις. Αυτή η εκχώρηση δεν συμπεριλήφθηκε στις ε, συμφωνίες. Εξ ονόματος των αλλιέων του Σεν Φιέκο Μισελόν, μία επισημοποίηση αυτής της ε, συμφωνίας που θα μπορούσε να γίνει με απλό ταχυδρομείο. Αυτή τη στιγμή οι συμφωνίες αυτές θα έχουν οριστικοποιηθεί. Θα μπορούσε η κυρία Επίτροπος να μας κάνει κάποιες διευκρινήσεις για το θέμα αυτό. Ο κύριος Φερέιρα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Οι πολυμερείς συμφωνίες, τα διεθνή υδατά θα οδηγήσουν στη βιωσιμότητα των αλλιευμάτων διαχρονικά. Θα πρέπει να έχουμε ε, συστημική προσέγγιση ως προς τη διατήρηση των αλλιευτικών πόρων, έτσι ώστε να εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο. Γι' αυτό θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα κενά που υπάρχουν στο σύστημα επιθεώρησης, ιδιαίτερα ως προς την παράνομη αλίευση. Υπάρχουν ε, μεγαλύτερες απαιτήσεις στα κράτη-μέλη και μέσα στα πλαίσια της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, καθώς και της ε, πολυμερούς συμφωνίας. Αυτό δεν θα πρέπει να το αγνοεί η Επιτροπή. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τα μέσα επιτήρησης και επιθεώρησης. Αυτό σημαίνει περαιτέρω χρηματοδότηση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας μέσα στα πλαίσια των νομικών βάσεων που διαθέτουμε στα πλαίσια της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και τη μέγιστη χρηματοδότηση που προβλέπεται στην περίπτωση με τις τάξεις του 50%. Σούπερ για ένα λεπτό. Danke, Herr Präsident. Auf der Jahrestagung der στην συνεδρίαση της ε, ΝΑΦΟ έγινε μια τροποποίηση της παλαιότερης ε, σύμβασης και θα πρέπει να διευθυνθούμε γιατί. Είναι σημαντικό να δούμε γιατί η βέλτιστη εκμετάλλευση των αλληλευτικών αποθεμάτων χρειάζεται ένα βιώσιμο αλληλευτικό μοντέλο για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη διατροφή των μελλοντικών γενεών μέσα από τα ψάρια. Και για τι συμφωνίες αυτές θα πρέπει, στις συμφωνίες αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι μικρές αλληλευτικέ ομάδες, οι οικογένειε των αλλιέων μαζί με τις οικογένειές τους, οι οποίοι θα πρέπει να προστατευθούν από παράνομους στόλους λαθρέα αλίες με μεγάλα δίχτυα πολύ συχνά. Ε, ε, ναι, θα πρέπει να προωθήσουμε την αλλία, αλλά προστατεύοντας ταυτόχρονα τις ε, μικρές, ε, τη μικρή βιο... την αλία μικρής κλίμακος, ούτως ώστε να είμαστε πιο βιώσιμοι μελλοντικά, να ασκήσουμε μια πιο βιώσιμη ελευτική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να κλείσουμε τη συζήτηση, πρώτα η ξενόμενη τη Επιτροπής, η κυρία Δαμανάκη, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητές για τη θαυμάσια δουλειά τους. Και θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω και όλους τους παρεμβαίνοντες για τα σχόλιά τους. Κατανοώ ότι πρόκειται για πολύ σημαντικές εκθέσεις, διότι μετά από αυτές τις τροποποιήσεις βελτιώνεται δραστικά η κατάσταση. Ειδικότερα έχουμε βελτίωση της του μηχανισμό ελέγχου και τις στάσεις μας γενικά όσον αφορά την παράνομη αλληλεία. Η παράνομη αλληλεία, συμφωνώ με όλους, ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά, διότι καταστρέφει τη βιωσιμότητα των πόρων και είναι απειλή για τις παράκτιες κοινότητές μας. Διότι αν καταρρεύσουν αυτοί οι πόροι, μετά οι παράκτιες κοινότητές μας δεν έχουν κανένα μέλλον. Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε αυτά τα συστήματα ελέγχου και οι τροποποιήσεις, οι τροπολογίες, μεταρρυθμίσεις αν θέλετε αυτών των προσεγγίσεων μας βοηθούν ακόμη. Χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους και ενδεχομένως περισσότερη χρηματοδότηση για να εφαρμόσουμε σωστά αυτούς τους κανόνες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν είναι εύκολη υπόθεση το να αντιμετωπίσουμε σωστά την κρίση. Εν πάση περιπτώσει θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχω ένα τελευταίο σχόλιο. Θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε σχέση με τη διαδικασία συναπόφασης μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωκοινοβουλίου και Κομισιόν. Αν θελήσουμε να ε, τροποποιήσουμε τις αποφάσεις RFMO και να τις μεταγράψουμε. Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ με την άποψη ότι αυτές οι πόδα περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης αλληλείας είναι πολύ σημαντικές για την πολιτική μας και πρέπει να προωθήσουμε την δραστηριότητά τους για να προωθήσουμε την νόμιμη αλληλεία παγκόσμια. Ακόμη, αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε να γίνει η σωστή εφαρμογή των αρχών μας παγκοσμίως, τότε η βιωσιμότητα της αλληλείας εξασφαλίζεται. Ακόμη, καλωσορίζω όλες τις προτάσεις σε σχέση με το πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τη συνεργασία. Καλωσορίζω και την πρόταση για την δημιουργία ενός παγκοσμίου μητρώου αλληλευτικών σκαφών. Ε, πρέπει όμως να γίνουν πολλά πριν φτάσουμε εκεί. Αν θέλουμε λοιπόν πραγματικά να προχωρήσουμε και να ενισχύσουμε αυτή τη διεθνή συνεργασία χρειάζεται να επισπεύσουμε την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται σε αυτές τις οργανώσεις. Γι' αυτό η Κομισιόν ζητάει περισσότερη εκχωρήση αρμοδιοτήτων. Βεβαίω και σεβόμαστε την διαδικασία συναπόφαση. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ένα νέο περιβάλλον τώρα και κατανοούμε ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφασίζουν για την εκχώρηση εξουσιών προς εμάς. Παρόλα αυτά όμως υπογραμμίζω ότι δεν είναι το πρόβλημα μόνο υπόθεση της Κομισιόν. Μιλάμε για τη διεθνή φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή διακυβεύεται όταν καθυστερούμε τη μεταγραφή των αποφάσεων των πόδα. Γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει να πετύχουμε μια καλύτερη ισορροπία. Χρειαζόμαστε ισορροπία. Συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα. Πρέπει να βελτιωθεί όμως αυτή η ισορροπία και είμαι διαθέσιμη να συζητήσω με το Κοινοβούλιο πώς μπορούν τα μέτρα των πόντα να μεταγράφονται πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλέσσα για δύο λεπτά. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, chciałem podziękować wszystkim e, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή φάνηκε ότι όλοι συμφωνούμε. Οι τροπολογίες οι οποίες ε, εισήχθησαν ήταν αναγκαίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φράγκα που πραγματικά έκανα αυτό το έργο της Επιτροπής. Αλλά καταρχήν θα ήθελα, πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς κυρία Επίτροπε, γιατί ήταν μεγάλη χαρά η συνεργασία μαζί σας. Ε, βλέπω ότι κατανοείτε καλά την δυναμική διάσταση ε, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Και στην περίπτωση αυτή, οι τροπολογίες, που αφορούν τις τροπολογίες στη Σύμβαση, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτές τις αλλαγές και να τις στηρίξω. Στο εξή νομίζω ότι η συμφωνία μας στον αφορά τις διαπραγματεύσεις θα προχωρήσει, θα γίνει με έναν ταχύ ή τρόπο χωρίς ε, τριβές και ιδιαίτερος με ψηλό επίπεδο διαφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις συνεργασίες σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να πω στην Επίτροπε ότι όσον αφορά τον τελευταίο αυτό κανονισμό της ΝΕΑΦΚΑ που θα εγκρίνουμε αύριο. Δεν είναι ένα καλό παράδειγμα, γιατί αυτό το οποίο συνέβη είναι αυτό το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Αυτή την πρόταση η Επιτροπή την παρουσίασε πολύ αργά. Στη συνέχεια άλλαξε τη διαδικασία. Από μια διαβούλευση περάσαμε σε μια διαδικασία συναπόφασης και η πρόταση στο σύνολό της τελικά είναι ε, σύμφωνα με, με τη συμβαστική αυτή λύση αποφεύγουμε το άρθρο 48 του κανονισμού που είναι αυτό το οποίο προβλέπει την τροποποίηση αυτού του κανονισμού για το μέλλον ούτως ώστε να μεταγραφεί σε κοινοτικό κανονισμό ε, να μεταγραφούν οι, οι, οι διάφορες συστάσεις. Και ακριβώς ε, υπάρχουν ε, κάποιες κατεξουσιαστικές πράξεις που περνούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι διατηρήσαμε τη διαδικασία συναπόφαση και υπάρχει μια σημαντική, ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά τη σωστή λειτουργία. Κυρία Επίτροπε, εγώ δεσμεύομαι εδώ δημόσια, ούτω ώστε στο μέλλον να μην ε, εμποδιζόμαστε στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, υποχρεώσεων μας. Θεωρώ ότι ως σημείο κίνησης αυτός ο συμβιβασμός συνιστά μια πρόοδο και θεωρώ ότι η Επιτροπή θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει σωστά τις νέες αυτές αρμοδιότητες που τις εκχωρούν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε ε, και είμαι βέβαιη ότι τα πράγματα μελλοντικά θα λειτουργήσουν πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία συνάδελφη, κυρία Επίτροπε. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 12.30. Η μερίσια διάταξη προβλέπει τώρα τις ε, παρεμβάσεις ενός ε, λεπτού ε, και συνάδελφοι θα διακόψουμε για ένα λεπτό περίπου για να ετοιμαστεί η συζήτηση των παρεμβάσεων όχι πάνω από ένα λεπτό. Οπότε όσοι θέλετε ή έχετε παρέμβαση παραμένετε, οι υπόλοιποι μπορείτε να αποχωρήσετε.